das protokoll und die 10ης ε, ε, Σεπτεμβρίου είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων